ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου έχει τη διάθεση του το Κοινοβούλιο. Τα πρακτικά του, της συνεδρίασης θα υποβληθούν ε, στην επόμενη ημέρα της ονομέλειας για έγκριση. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε έτσι τις εργασίες